φορά που επιβάλλουμε κυρώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για αυτό το θέμα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη που είναι οι παρεμβάσει ενός λεπτού. Έχουν ζητήσει διάφοροι το λόγο για να παρεύουν. Ο κύριος Ζαζάντα πρώτα. Ε, ένα λεπτό, έτσι, οι παρεμβάσεις ενός λεπτού υπενθυμίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηρες ε, μητέρες και οι δικαιωμένοι στα ευρωπαϊκά αεροδρομία. Ο κανονισμός 11-2007 ορίζει πως ε, οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να βοηθούνται στα αεροδρόμια, αλλά συχνά δεν γίνονται σεβαστές οι διατάξεις ε, αυτές. Παραδείγματος χάρη, σε κάποια πλάνα τα οποία προετοίμασε η Κομισιόν βλέπουμε μητέρες με μικρά παιδιά που δεν ε, γνωρίζουν καν ότι δικαιούνται βοήθεια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει το όνομα του κανονισμού και να πούμε πως ισχύει και για γονείς που ταξιδεύουν με τα παιδιά τους. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη για τους πολίτες μας. Κύριε, Κύριε αυτό το λόγο. Είμαι μέλος στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ως Ισπανίδα και Ευρωπαία πολίτης και ως θύμα της τρομοκρατίας από τότε που η ΕΤΑ ε, δολοφόνησε τον αδερφό μου στη Σεβίλη, απευθύνομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταγγείλω την κυβέρνηση της Βενεζουέλα και τον πρόεδρό της που επέτρεψε τρομοκράτες της ΕΤΑ να πάνε και να εκπαιδευτούν εκεί, στο εδαφό της, στην επικράτειά της. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για τον Τσάβε στην κυβέρνησή του παρόλο που υπάρχει εναντίον τους καταδίκη. Υπάρχει μεγάλη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πλήττεται έτσι η ασφάλεια οποιοδήποτε Ευρωπαίου πολίτη. Απαιτώ λοιπόν από την Ισπανική κυβέρνηση να αναλάβει δράση για αυτή τη μεγάλη ταπείνωση την οποία εφίστανται όλοι οι Ισπανοί. Ο Σαπατέρο δεν είναι δυνατόν να στοιχίζει να σιωπά, ενώ ο πρέσβη ε, τη Βενεζουέλα ε, συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να υπάρξει μια δράση με θάρρος από πλευράς της Ισπανικής κυβέρνησης κατά της ΕΤΑ. Η συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στις ΕΤΑ και τους ΦΑΡΚΕ είναι ένα άλλο θέμα. Πάλι στο έδαφος της Βενεζουέλας με τον δικαστή Βελάκο, όπως ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν η Ισπανική κυβέρνηση να δίνει το χέρι στον Τσάβες, ο οποίος κάνει την Βενεζουέλα καταφύγιο για τρομοκράτες. Ο πρόεδρος μιας χώρας σαν την Ισπανία, όπου η τρομοκρατία ε, μας έχει πονέσει τόσο πολύ, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει να αγνοεί αυτό το πρόβλημα και θα έπρεπε να δώσει μία απάντηση αυτή που αξίζει οποιοδήποτε πολίτης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χιμένεθ, αλλά ε, να σας πω ότι έχουμε ένα λεπτό για τον καθένα. Η κυρία Στήλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να σας πω ότι στις 18 ε, Οκτωβρίου πολλοί συνάδελφοι, 36 μέλη, ε, βραβεύτηκαν από, την Ευρωπαϊκή, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνευμόνων ε, για την προσπάθειά τους όσον αφορά την καταπολέμηση, την αντικαπνιστική τους δράση και όσον αφορά τον έλεγχο των ε, ε, καπνοβιομηχανιών. Μονάχα 10 από τις 27 χώρες μέλη έχουν ε, αυτή τη στιγμή πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και επομένως ζητούμε και από τις υπόλοιπες χώρες άμεσα να προχωρήσουν σε μια τέτοια αντικαπνιστική δράση. Έχουμε διαπιστώσει ότι στις ε, χώρες όπου έχει εφαρμοστεί αυτός ο πλήρης αντικαπνιστικός νόμος έχουμε 18% λιγότερα παιδιά τα οποία φτάνουν στα νοσοκομεία με αναπνευστικά ε, προβλήματα. Αυτά με την ευκαιρία της βράβευσης 18 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίντερς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την ψηφοφορία της προηγούμενης εβδομάδας της ε, Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού να παγώσει μισθούς ε, και επιδόματα των επιτρόπων εάν δεν αλλάξει ο κώδικας συμπεριφοράς για να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως του κυρίου Μακρύβη ο οποίος ερευνάται για πιθανά συγκρουόμενα συμφέροντα. 200 αιτήματα έγιναν για το τι κάνουν οι επίτροποι, για να λάβουν οι επίτροποι άλλα καθήκοντα μετά τα καθήκοντά του στου και μόνο ένα απορρίφθηκε. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει πολύ ευρεία και χαλαρή ερμηνεία. Κύριος Κόσλικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή κυβέρνηση της Σλοβακίας προτείνει πράξεις οι οποίες μειώνουν την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Η πρόταση για να γίνουν αλλαγές στο Σύνταγμα προς αυτή την κατεύθυνση υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο χωρίς προηγουμένως να γίνει διαβούλευση. Στην Σλοβακία λοιπόν παραμορφώνεται η δημοκρατία σήμερα. Υπάρχει και ένα άλλο γεγονός ότι ο επικεφαλής του του Δικαστηρίου αποκλείστηκε δύο φορές από το Κοινοβούλιο όταν συζητούσαμε τις νέες πράξεις για το δικαστικό σώμα. Είναι λοιπόν αυτή η πράξη περιορίζει και τον αριθμό των δικαστών στο Δικαστικό Συμβούλιο πριν λήξει η θητεία τους και αυξάνει τον αριθμό των πολιτικών διορισμών στην Επιτροπή που διαλέγει τους δικαστές. Αυτή είναι μια μικρή μόνο εικόνα για το τι κάνει η κυβέρνηση στη Σλοβακία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόγκος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα σήμερα για την Ουγγαρία. Πριν από πάνω από 150 χρόνια πριν ε, οι Ούγγροι πατριώτες ε, πήραν τα όπλα για να παλέψουν για την ελευθερία, την ισότητα και την ε, αδελφοσύνη. Οι 13 επικεφαλής στρατηγοί της αποτυχημένης επανάστασης εκτελέστηκαν σε μια πόλη που σήμερα βρίσκεται στην Ρουμανία. Όμως το 1956 ξανά εκδηλώθηκε η επιθυμία μας για ελευθερία αυτή τη φορά από τον κομμουνισμό. Οι 13 λοιπόν μάρτυρες, από τους μάρτυρες αυτούς μόνο τρεις ήταν Ούγγροι, κάτι το οποίο βεβαίως αποδεικνύει το ότι η ελευθερία είναι κάτι το πανανθρώπινο και βεβαίως τιμά και την αλληλεγγύη των ε, εθνών. Ο κύριος Δίας Δεμέρα Γκαρθία Κονσουέγρα. Ευχαριστώ. Εδώ θέλω να καταδικάσω τη συμπεριφορά του Τσάβες που παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο συνάδελφος Τουργάης το Καράκας συνελήφθη. Είναι η πρώτη φορά που τα βάζει με ένα μέλος του ΕΛΚΑ η κυβέρνηση του Τσάβες. Εμείς ως ευρωβουλευτές καταδικάζουμε τη συμπεριφορά αυτή πρέπει να επενθυμίσουμε τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχέ όπω είναι η ελευθερία, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά βέβαια τέτοια πράγματα δεν αρέσουν σε αυτούς που θέλουν να επιβάλλουν ολοκληρωτικές ιδέες. Ελπίζουμε όμως ότι θα υπάρξει αντίδραση από την ε, αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα. Τι μπορούμε να περιμένουμε όταν προστατεύει τον ε, Τόκερ που είναι ε, τρομοκράτης που είναι από τους δολοφόνους της ΣΕΤΑ και έχει βρει κατεφύγιο στην επικράτεια της Βενεζουέλας πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε από τον Τσάβες να δώσει δικαιοσύνη. Τίποτα. Τέτοιες συμπεριφορές κυρία Πρόεδρε αξίζουν δράση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την δικιά μας αποστροφή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταμπάτζη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε πως ε, ο διαχωρισμός Γερμανίας καταδείκνει το παράλογο του διπολισμού και βεβαίως η επανένωση Γερμανίας ήταν προϋπόθεση για την επανένωση ολόκληρη Ευρώπη. Κάτι το οποίο νιώθαμε και εμεί στην Ουγγαρία. Η επανένωση λοιπόν τη Γερμανία αποτέλεσε την αρχή τη επανένωση τη Ευρώπη. Η πτώση του τείχου του Βερολίνου τερμάτισε το διχασμό στη μεταπολεμική Ευρώπη και ως Ούγγρος είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τους Ούγγρους ηγέτες και πολιτικούς που είχαν τότε το θάρρος να ανοίξουν τα σύνορα με την Αυστρία για δεκάδες χιλιάδες ε, Ανατολικογερμανούς αγνοώντας την συνθήκη που είχαν υπογράψει με την Ανατολική Γερμανία και έριξαν έτσι το πρώτο τούβλο αν θέλετε αυτό το τείχος του Βερολίνου. Γιούλα Χόρνο, Υπουργός Εξωτερικών έκανε μία ιστορική πράξη. Σας ευχαριστώ κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μόλις επέστρεψα από την Ισλανδία μετά από την πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και στη διμερή αυτή επίσκεψη είχαμε πολύ ενημερωτικές συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της Ισλανδίας ε, όσον αφορά την αίτησή τους. Όταν συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Αλληλείας έθιξα την σημαντική αύξηση του επιτρεπόμενου συνολικού αλλιεύματος σκουμπριού. Ειδικά ε, για αυτό το ψάρι. Και με ικανοποίηση μείωσα από στις 12 Οκτωβρίου στο Λονδίνο η Ισλανδία θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα άλλα κράτη που βρέχονται από τη Βόρεια Θάλασσα και ελπίζω να καταλήξουμε σε μία λύση. Εξακολουθεί βεβαίως να είναι πάρα πολύ, ε, να είναι έντονες συνέπειες της κρίσης στην Ισλανδία, γι' αυτό θα πρέπει επίσης να υπάρξουν και διαπραγματεύσεις για την τράπεζα iSave με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία για να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κουμουτσάκος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο επίτροπο ε, κύριος Μπαρνιέ είναι παρόν σήμερα εδώ, καθώ το θέμα στο οποίο θα αναφερθώ γνωρίζω ότι τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Οι φυσικέ καταστροφέ έχουν ανυπολόγιστο κόστο σε ανθρώπινε ζωέ και οικονομικέ υποδομέ. Η αντιμετώπιση του είναι κοινή πρόκληση και απαιτεί κοινέ δράσει είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη η ευρωπαϊκή ένωση να μπορεί να απαντά αποτελεσματικά σε τέτοιε καταστάσει έκτακτη ανάγκη. για να το πετύχει η ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει καλύτερα τι δυνατότητε που έχει αλλά και να κινητοποιήσει του ευρωπαίου πολίτε. η μακρά ευρωπαϊκή παράδοση του εθελοντισμού και η αρχή τη αλληλεγγύη δίνουν στέρεη βάση για να το πετύχουμε. ήρθε λοιπόν η ώρα για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού σώματο εθελοντών όπω ακριβώ προβλέπει το άρθρο 214 παράγραφο 5 της συνθήκης Λισαβόνα. Υπενθυμίζω μάλιστα ότι το 2011 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών θα ενισχύσει το ρόλο και την εικόνα της Ευρώπης και θα κερδίσει το μυαλό και την καρδιά των Ευρωπαίων αλλά και των πολιτών όλου του κόσμου. Το κοινοβούλιο μας έχει χρέος να δραστηριοποιηθεί επιγόντως για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών. Ο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα στη χώρα μου. Θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να ε, γίνουν οι απαραίτητοι σχεδιασμοί έτσι ώστε να μειωθούν ε, οι εκπομπές ε, κυρίως ε, όσον αφορά δε όσον αφορά το, το τσιμέντο, παραγωγή τσιμέντου πρέπει να πω ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα γιατί έχει υπολογιστεί ότι βάσει των νέων αρχών μείωση διοξιδίων του άνθρακος θα έχουμε αύξηση της τιμής του τσιμέντου κατά περίπου 30%. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί ε, χώρες οι οποίες δεν μπορούν να ακολουθήσουν το γρήγορο βήμα της Γερμανίας ή της ε, Γαλλίας θα πρέπει να ε, βοηθηθούν. Η κατάσταση αυτή οδηγεί και σε, ένα άλλο, σε μια άλλη επίπτωση. Μερικοί κατασκευαστές και μερικοί παραγωγοί θα αναγκαστούν να φύγουν εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Το αντιδημοκρατικό ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης χθες 5 Οκτώβρη ταυτίζει τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες με τον εξτρεμισμό στο όνομα της καταπολέμησης του εξτρεμισμού προτείνει τον περιορισμό και την κατάργηση βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση τα δικαιώματα του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε ακόμη και την απαγόρευση δράσης πολιτικών κομμάτων ιδιαίτερη αναφορά επιφυλάσσει το κατάπτυστο αυτό ψήφισμα μπορείτε να μιλάτε με λίγο, ρυθμό γιατί ήδη μπορούν να ακολουθήσουν Στο αυτό ψήφισμα για την Ελλάδα και τους μεγάλους εργατικούς λαϊκούς αγώνες που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα ενάντια στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης στη χώρα μας καθώς και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ταξική πάλι δεν σταματάει με αντιδραστικά ψηφίσματα και νόμους. αποτελεί κινητήριο μοχλό της ιστορίας αναπόφευκτο προϊόν του συστήματος γέννημα της βαρβαρότητας της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. η πάλι της εργατικής τάξης η ανασυγκρότηση και αντεπίθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος σε ολόκληρη την ευρώπη μπορεί να τοποθετήσει τα ψηφίσματα αυτά εκεί που ανήκουν στα σκουπίδια της ιστορίας το κομμουνιστικό κόμμα ελλάδας καλεί την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να καταδικάσουν έμπρακτα το αντιδραστικό ψήφισμα με την ένταση της πάλης τους ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου της ευρωπαϊκής ένωσης των αστικών κυβερνήσεων δυναμώνοντας την προσπάθεια για την οικοδόμηση της κοινωνικοπολιτικής συμμαχίας της εργατικής τάξης αυτοαποσχολούμενων που θα διεκδικήσουν αλλαγές προς όφελος του λαού. Ευχαριστούμε. Η κυρία Αντρικάιν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα στις Βρυξέλλες γίνεται διάσκεψη κορυφής ε, Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κλίμα, το εμπόριο είναι πράγματα που είναι στην ημερήσια διάταξη, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα <coughs> και η θανατική ποινή και τα στρατόπεδα εργασίας. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα. Θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι άλλο σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που είναι το Θιβέτ. Λυπούμεθα που ο διάλογος ανάμεσα στο Δαλάι Λάμα και τις κινέζικες αρχές πηγαίνει πάρα πολύ αργά. Ο τελευταίος γύρος έλαβε χώρα τον αύριο που μας πέρασε. Οι συναντήσεις είναι εντελώς ποραδικές και καταστρέφονται ουσιαστικά από την έλλειψη εμπιστοσύνη που επικρατεί. Ο Δαλάι Λάμα έχει ήδη πει ότι δεν θέλει αυτονομία, θέλει περισσότερη αυτοδιάθεση. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει διάλογος και να αποφύγουμε τη βία. Το διάλογο το θέλει ο Δαλαϊδλάμα και θα κάνει ό,τι μπορεί για να το διευκολύνει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαντίμ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε στην Ρουμανία αυτή τη στιγμή ε, υποφέρουμε από ε, μεγάλη λογοκρισία. Ε, το NCA, το Εθνικό Συμβούλιο για τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα λογοκρίνει ακόμα και τον Θερβάντες και τον Γκέτε και άλλους γνωστούς συναδέλφους και συγγραφείς, συγγνώμη αυτή τη στιγμή ανεξάρτητη τηλεοπτικοί σταθμοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν ε, και ε, ε, αισθανόμαστε ότι όλη η χώρα και όλη η πολιτιστική παραγωγή είναι ένα νεκροταφείο από το οποίο βγαίνουν ζόμπι που λογοκρίνουν την αλήθεια. Θέλουμε να μας βοηθήσετε να κερδίσουμε, να πάρουμε πίσω αυτά που είχαμε κερδίσει με τους αγώνες της προηγούμενους της δεκαετίας. Άρκιν, η κυρία Άρκιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νωρίτερα απόψε ακούσαμε για τις ε, κοινωνικέ διατάξει τη συνθήκη Λισαβόνα που υποχρεώνουν την Κομισιό να λάβει υπόψη στις κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεων. Το έχει κάνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις όταν επιμένει πως θα πρέπει μέχρι το 2014 να συμμορφωθεί με το Σύμφωνο σταθερότητα η Ιρλανδία. Ναι, εντάξει. Οπωσδήποτε η εξυγίανση των οικονομικών είναι σημαντική, αλλά έχουμε την εντύπωση πώ μόνο αυτό μετράει. 3% μέχρι το 2014, Αλλιώ. αυτό δηλαδή ότι μας λένε οι Βρυξέλλες πριν, μας είπαν από την Βουλική Προεδρία πως δεν είναι απαραίτητη η λιτότητα χωρίς αύριο. Κι όμως αυτό ακριβώς αντιμετωπίζουμε. Ναι, χρειάζεται να ξαναφτάσουμε στο 3% αλλά χρειάζεται ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Αποδέχομαι πως πολλές από τις δυσκολίε τις έχουμε προκαλέσει εμείς. Αλλά αν δεν σκεφτούμε λίγο παραπέρα από την λιτότητα θα οδηγηθούμε σε πολύ χειρότερα. Και ακόμα τέσσερις επιχειρήσεις κλείνουν την ημέρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Σας ευχαριστώ. Τον, κύριο, τον λόγο έχει η κυρία Κρίτζολφσκα. Ευχαριστώ. Πρόσφατα στην Πολωνία αντιμετωπίσαμε περιπτώσεις ψυχοτρόπων ε, ουσιών, ανθρώπων δηλαδή που χρησιμοποιούσαν ψυχοτροπικές ουσίες που οδήγησαν σε θάνατο. Δεν υπάρχουν σωστοί κανονισμοί, κατάλληλοι κανονισμοί, έτσι ώστε οι αρχές να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών. Οι χρήστες δε των ψυχοτροπικών ουσιών πιστεύουν ότι εφόσον δεν απαγορεύονται, δεν κάνουν και κακό. Όμως οι ουσίες αυτές πολλές φορές είναι περισσότερο βλαβερές από ό,τι τα ναρκωτικά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτές οι ουσίες και κυκλοφορούν ε, έτσι, πρέπει να φροντίσουμε εμείς να πάρουμε μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι θα έπρεπε να φροντίσει για μέτρα ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για τις επιπτώσεις και τις παρενέργειες που μπορεί να έχουν οι ψυχοτρόπες ουσίες. Ευχαριστώ κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ. Όπως είπαν σήμερα οι Financial Times, ε, η Επίτροπος Έρευνας είπε πως θα υπάρχει έλλειψη στην Ευρώπη όσον αφορά την έρευνα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την έρευνα στον ιδιωτικό τομέα με επιχειρηματικά κεφάλαια και οικονομικές πρωτοβουλίες. Όμως οι προτάσεις της Ένωσης για να μην επαναληφθεί η χρηματοπιστωτική χρήση βάζει το επιχειρηματικό κεφάλαιο μαζί με τους κερδοσκόπους όπως τα hedge funds στο ίδιο καλάθι. Ενώ ξέρουμε πως αυτά τα κεφάλαια βοηθούν μικρές επιχειρήσεις που ξεκινούν για να κυριαρχήσουν μετά στην παγκόσμια οικονομία όπως το Google, το Facebook και το Skype. Και συχνά έχουν την εμπειρία και την πρόσβαση στην αγορά, ε, τις επενδύσεις που χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσει σε μια περίοδο τριών μέχρι 7 ετών. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ και στη Ιαπωνία και τέλος πρέπει να ακούσουμε τα όσα είπε βεβαίω και η Επιτροπός Έρευνας. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Αλφανό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ να πω στο Κοινοβούλιο ότι στην προηγούμενη Κυριακή στην επίσκεψη του Πάπα ε, στο ε, Παλέρμο ε, δεν εφαρμόστηκε ή δεν εφαρμόστηκαν οι αρχές της προστασίας της έκφρασης, ελευθερίας έκφρασης. Υπήρχε μία μια επιγραφή που έλεγε ότι το σπίτι μου είναι το σπίτι της προσευχής αλλά εσείς το καταλεηλατίσατε. Ε, και υπήρχε και ένα άλλο, μια άλλη ε, ταμπέλα που έλεγε I love billing. Ε, νομίζουμε ότι αυτού του είδους η άσκηση δύναμης από τις αστυνομικές δυνάμεις καταλύουν το δημοκρατικό κράτος και την ελευθεροτυπία καθώς επίσης και την ελευθερία έκφρασης ενώ ο πρόεδρος, ενώ ο πρωθυπουργός Μπερλουσκόνη μπορεί να βλασφημεί ε, χωρίς κανένα πρόβλημα, ε, δεν είναι δυνατόν, ε, δεν επιτρέπεται στον απλό κόσμο να εκφράζει την άποψή του. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό, το, οποίο, το κενό που υπάρχει ανάμεσα στο, στον κόσμο και στις, στα θεσμικά όργανα και τους θεσμούς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στενάσκο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, παρά τα μέτρα καταπολέμησης της ε, κρίσης, ε, διαδηλώσεις και απεργίες δείχνουν πως η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Δυστυχώς ε, τα μέτρα αυτά με τα οποία προσπαθούν οι κυβερνήσεις να μπαλώσουν τις τρύπες του προϋπολογισμού και να ξεπληρώσουν τα δάνεια δημιουργούν νέα κρίση με το να μειώνουν το εισόδημα και την ποιότητα ζωή των πολιτών. Ίσως έχει φτάσει η ώρα να αλλάξουμε σκοπό και να βάλουμε πρώτα απ' όλα το συμφέρον των πολιτών που συνεχώς φτωχαίνουν πάνω από το συμφέρον των τραπεζών οι οποίες εξακολουθούν κατά μυστήριο τρόπο να αυξάνουν το κέρδη τους. Εάν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να χάσει κάποιο από αυτή την υπόθεση, δεν θα πρέπει να είναι πάντα ο κοινό πολίτη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ για τη Βενεζουέλα θα μιλήσω, γιατί δεν είναι δημοκρατία μόνο ερχόμαστε και να ψηφίζουμε. Είναι να νιώθουμε ασφάλεια, ισότητα και να ζούμε σε ένα καθεστώς ελευθεριών, όπου και η ιδιωτική περιουσία πρέπει να τύχεται σεβασμού. Ενώ ένα σωρό επιχειρήσει στη Βενεζουέλα απειλούνται. Υπάρχει μια επιχείρηση που φτιάχτηκε από Ισπανούς από τα Κανάρια νησιά. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Την έχουν πάρει όμως τη Βενεζουέλα, όπως και πολλές άλλες που μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών τελικά ε, καίγεται και τους την παίρνουν. Χτες πήραν γη. Ε, παλιότερα. Σήμερα παίρνουν επιχειρήσεις. Οι πολίτες δεν νιώθουν ελεύθεροι. Οι επιχειρηματίε νιώθουν να απειλούνται η Βενεζουέλα θα έπρεπε να είναι αυθεντική δημοκρατία και όχι να βρίσκουν εκεί καταφύγιο τρομοκράτες. Ευχαριστώ. Ρενιέ τώρα, παρακαλώ. Η κυρία Ρενιέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην εβδομάδα δράσης της ε, Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένους Μεταφορές που λαμβάνει χώρα αυτή την εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Αφορμή για αυτό ήταν η επιθετική πρακτική μιας παγκόσμιας εταιρείας κατά των υπαλλήλων τους οι οποίοι θέλησαν να συνδικαλιστούν. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο δεν έχει φτάσει ακόμα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και βέβαια αυτό το εκμεταλλεύονται οι εταιρείες. Σύμφωνα με το τουρκικό εργατικό δίκαιο ένα συνδικάτο μπορεί να δημιουργηθεί σε μια εταιρεία εάν φτάσει ένα ποσοστό πάνω από 50% των εργαζομένων. Η UPS λοιπόν με σκληρό τρόπο σταμάτησε την οργάνωση των ε, εργαζομένων. Απέλησε άμεσα 175 άτομα που προσπάθησαν να συνδικαλιστούν και ζήτησαν να αναγνωριστεί το συνδικάτο, το συνδικάτο τους. Σταμάτησαν λοιπόν την εργασία οι συναδελφοί τους. Με τον φιλικό αυτό προς επιχειρήσεις νόμο θα δημιουργηθεί στην Τουρκία ένας χώρος που δεν θα έχει καθόλου συνδικάτα. Σας ευχαριστώ κυρία Μπιλμπά Παραντικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. 18 Οκτωβρίου ξεκινάει στο Γιαρκαβίρ στην Τουρκία μια δίκη κατά 18 ε, πολιτών. 14 έχουν εκλεγεί, δύο δήμαρχοι και δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Κατηγορούνται ότι ειρηνικά υποστήριξαν τις πολιτικές τους θέσεις και μπορεί να έχουν 15 χρόνια ποινή φυλάκισης. Οι κρατήσεις αυτές και οι φυλακίσεις αυτές είναι ένα παράδειγμα μόνο από τόσα υποφέρει η κουρδική μειονότητα στην Τουρκία. Το Φεβρουάριο είχαμε αποφασίσει ότι θα αναλύσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χώρα αυτή για να δούμε αν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Εμεί πιστεύουμε ότι η πρόοδο δεν είναι αρκετή. Πρέπει να στηρίξουμε κάθε κίνημα αλληλεγγύη προ το κουρδικό κίνημα τη Τουρκία. Θέλω να ζητήσω από το Κοινοβούλιο να στείλει επίσημη αντιπροσωπεία στον Τικιαρκαβίλ, στην δίκη αυτή δηλαδή, για να παρακολουθήσει τη δίκη. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλβάου, Η κυρία Κρετή έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι που μπορεί να συμβεί στη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης ε, είναι ότι ε, μπορεί τελικά ε, να προκύψει και πολιτική κρίση. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μου η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει ανήκουστα μέτρα λιτότητας και πρωτοφανή μέτρα ε, ε λιτότητας που έχουν οδηγήσει τον κόσμο στον ε, στο να ζει χωρίς θέρμανση, χωρίς φάρμακα, χωρίς περίθαλψη γιατί έχουν μειωθεί ε, στο μέγιστο βαθμό τα εισοδήματά τους. Ε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως έχουμε επίσης και φαινόμενα λογοκρισίας ε, και απαγόρευσης της ελευθερίας έκφρασης. Πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα δει από κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν ε, να αφήσουμε τη Ρουμανία να προχωρεί προς αντιδημοκρατικό δρόμο. Ευχαριστώ η κυρία Καρβάγιο.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 να αναφερθώ εδώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην ε, έκθεση που κάνει σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών σε επαγγέλματα υγείας. Εγώ καταδικάζω την έκθεση αυτή. Είναι μια ανάμιξη στην κυριαρχία των κρατών μελών. Παραβιάζει την επικουρικότητα και το θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία και στην ε, ελευθερία θρησκείας. Μιλάει για τις γυναίκες, για την άμβλωση, για την τεχνητή γονιμοποίηση και για την στήρωση. Μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο μικραίνουμε τη ζωή ασθενών που πάσχουν από ανίατες ασθένειες. Και λέει ότι όσοι δουλεύουν στην υγεία πρέπει να προσφέρουν ε, τη δυνατότητα αυτή και να το κάνουν δηλαδή. Δεν είναι αποδεκτή για μας μια τέτοια ρύθμιση στην Ευρώπη. Αντιφαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ανεύθυνο να τα βάζουμε με την εξωτερική πολιτική της Ισπανίας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να μιλάμε για κατάρτιση τρομοκρατών στη Βενεζουέλα. Υπάρχει διάλογος, υπάρχει συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, αλλά τα πράγματα αυτά που λέτε γίνονται εκτός συνόρων της Ισπανίας. Στο διάλογο με τη Βενεζουέλα έχουν ζητηθεί συγκεκριμένα μέτρα. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές αλλά και τις διπλωματικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους που έχουν ήδη πετύχει αρκετά πράγματα και ο διάλογος έχει καρποφορήσει για τον περιορισμό της τρομοκρατία στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μονίθ και έτσι εδώ ολοκληρώνονται οι παρεμβάσει ενό λεπτού. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση της κυρίας Κάισερ για συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσοχάρια Αφρική και